105 η σύνοδος των πρόεδρων των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών μου είπε ότι δεν υπάρχουν καθόλου αντιρρήσεις σε σχέση με την ε, κατεξουσιοδότηση πράξης κατεξουσιοδότηση πράξη από την Επιτροπή Ίντα. Εάν μέσα σε 24 ώρες δεν υπάρξει ούτε μια πολιτική ομάδα ούτε τουλάχιστον 40 μέλη τα οποία θα γίνουν αντίρρηση στις επόμενες 24 ώρες θα θεωρηθεί ότι αυτή η σύσταση έχει εγκριθεί. Αλλιώ θα τεθεί σε ψηφοφορία. Και η σύσταση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σχέση με το